όχι, θα περάσουμε στη ψηφοφορία. Κύριε Ράνστορφ, για το ίδιο θέμα θέλετε το λόγο. Ναι, Πρόεδρε. Για το ίδιο θέμα. Γνωρίζω ότι το γραφείο Ζαχάροφ είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα.